από τις 20 Ιουλίου του 2009. Έλαβα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και των ε, ε, Ευρωπαίων Δημοκρατών καθώς και των Πρασίνων ε, της Ευρώπης για την Ευρώπη των Πολιτών μερικές μερικά ψηφίσματα σε σχέση με αλλαγές σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και ε, διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπίες, τα οποία θα επισυναφθούν στα σημερινά πρακτικά. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσει στάσεις για τις αλλαγές αυτές, θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένε. Έχετε λάβει τις προτάσεις για τις αλλαγές από τα διάφορα κόμματα, δεν πρόκειται να τις διαβάσω, μπορείτε να τις εξετάσετε. Μία άλλη πληροφορία. Ε, οι τελικές δικαστικές αρχές ζήτησαν την άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή Ρομπέρτο Φιόρε, Ιταλού Ευρωβουλευτή, για ένα θέμα που εκκρεμωδικεί στο δικαστήριο της Βιτσέντζας. Με βάση τον κανονισμό, το αίτημα αυτό θα παραπεμφθεί στη νομική επιτροπή που είναι αρμόδια καθήλη για τα θέματα αυτά. Επίσης, η αρμόδια καθήλη επιτροπή ε, μου έθεσε ένα ερώτημα για ψήφισμα δεύτερης ανάγνωσης που θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της